Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ξεκινούμε τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής μας στα μέσα της θητείας. Πρέπει να προχωρήσουμε στις διαδικασίες που προβλέπει η μερίσια διάταξη. Εκλογή των, του Προέδρου ή της Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Ξεκινώντας από τον πρώτο ή την πρώτη Αντιπρόεδρο και φτάνοντας τον την τέταρτη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την προσέλευσή τους και δίνω απευθείας το λόγο στον συνάδελφο Γιάννη για την αρχική πρόταση. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα εξ ονόματα του κόμματο τη ε, ομάδα του ΕΛΚ να προτείνω την Ειρηνή Ματσόνη. Σα παρακαλώ για ψήφο εμπιστοσύνη και την εκλογή τη. Σα ευχαριστώ πολύ. Ringrazio il collega Peter Iar. Ci sono altri candidati alla carica di Presidente della Commissione. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες για την Προεδρία της Επιτροπής. Εάν όχι, θα έλεγα να διαβοήσει να ψηφίσουμε τον Πρόεδρο. Ringrazio i colleghi. Ευχαριστώ τους συναδελφούς. Ευχαριστούμε για αυτή την ψηφοφορία. Προχωρούμε με τις υπόλοιπες ψηφοφορίες. για την θέση του πρώτου αντιπροέδρου ή της πρώτης αντιπροέδρου. Έχω λάβει την υποψηφιότητα της κυρίας Παλιαδέλη. Με συγχωρείτε, ένα έξτρα. Είναι Ένα πολύ ευχάριστο έξτρα εκτό προγράμματο. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Γιάρ και όλη την αντιπροσωπεία του ΕΛΚ για αυτό τον υπέροχο φορό τιμή. Ξεκινά έτσι με πολύ όμορφο τρόπο η νέα μου θητεία στην Προεδρία αυτή τη Επιτροπής. Συνεχίζουμε με το δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έλεγα υποψήφια για τη θέση της πρώτης αντιπροέδρου υποψηφιότητα της κυρίας Παλιαδέλη. Προς στιγμή. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Προτείνω να ψηφίσουμε διαβοής. Και για την κυρία Παλιαδέλη. Για τη θέση του δευτέρου αντιπροέδρου λάβαμε την υποψηφιότητα του κυρίου Μάγερ. Δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Σε αυτή την περίπτωση προτείνω να ψηφίσουμε διανάταση της χειρός. Διαβοής μάλλον εννοεί πρόεδρος. Και ο συνάδελφος Μέγερ λοιπόν διαβοής έχει εκλεγεί. Τρίτη υποψηφιότητα, τρίτος αντιπρόεδρος, ε, τρίτη αντιπρόεδρος. Υποψηφιότητα Τουργκάης. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Διαβοής. Εξελέγει λοιπόν και ο πρόεδρος Ιτουργκάης τέταρτη υποψηφιότητα η κυρία Βασέσκου. Έχει υποβάλει υποψηφιότητα. Υπάρχουν άλλες ε, προτάσεις. Όχι. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση Ψηφίζουμε διανάταση τη χειρό, δηλαδή διαβοής. Και η συνάδελφο Μπασέσκου λοιπόν έχει εκλεγεί. Ευχαριστώ τα μέλη τη Επιτροπής. Παρακαλώ τους αντιπροέδρους να έρθουν κοντά μου στο Προεδρείο. Η συνάδελφο Παλιαδέλη, ο κύριο Μέγερ, που απουσιάζει παρόλα αυτά, είχε ένα πρόβλημα ταξιδιωτικό. Ο κ. Στουργκάη και η κυρία Μπασίσκου. Ο συνάδελφος Μποστινάρου, ο κ. Σολαβράκος, έχουν ζητήσει συγγνώμη για την απουσία του σήμερα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Έχουμε συγκροτήσει την Επιτροπή μας. Ο συνάδελφος Γιάρ θέλει το λόγο. Äh, äh, Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τα νέα μέλη του Προεδρείου για την εκλογή τους. Σας εύχομαι πολύ απλά η καλή και καρποφόρα συνεργασία να συνεργιστεί, γιατί είναι η πιο σημαντική επιτροπή, η Επιτροπή Αναφορών, γιατί ε, είναι η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την επεξεργασία των ε, καταγγελιών των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχόμαστε λοιπόν από πλευρά μας ό,τι καλύτερο και νομίζω ότι ως Επιτροπή στο έργο σας αυτό θα σας βοηθήσουμε, θα σας υποβοηθήσουμε. Σας εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο και είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε πολύ επιτυχείς. Nessun altro δεν ζητά το λόγο κάποιος άλλος συνάδελφος. Ιδέουσες ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους. Θα συνοδεύσουν τη δέσμευσή μου ως Προεδρού να δώσω και να προσδώσω τον κεντρικό καθοριστικό ρόλο που έχει η Επιτροπή αυτή στη διεξαγωγή των εργασιών του σώματός μας, του Κοινοβουλίου και στην οικοδόμηση της Ευρώπης των λαών. Ελπίζω ότι σε αυτό το δεύτερο ήμιση της ε, κοινοβουλευτικής θητείας η πείρα των πρώτων δυόμιση ετών θα χρησιμεύσει ώστε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, ώστε να εξεύρουμε απαντήσεις πιο ικανοποιητικέ για τους συμπολίτες μας. Εύχομαι ότι θα φανώ άξια με την καθημερινή μου προσπάθεια της ε, ομόφωνης ε, συγκατάθεσης και εκλογής και επαφίεμαι και στην ομάδα των αντιπροέδρων που με μεγάλη χαρά υποδέχομαι κοντά μου γιατί ξέρω ότι θα προσφέρουν την καθοριστική στήριξη που χρειάζεται για την εκπλήρωση της αποστολής μου. Δεν προβλέπονται άλλες διαδικασίες για τη σημερινή συνεδρίαση, οπότε θα κηρύξω τη λήξη της συνεδρίασης ως την επόμενη συνάντηση που έχει οριστεί στο πρόγραμμά μας για τις 26 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Καλό σας απόγευμα.